in the future. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην ε, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας που έχει σήμερα την ευκαιρία να συζητήσει με τον Επίτροπο, τον κύριο Τόνιο Μπόργκ, το θέμα της σήμανσης ε, του κρέατος αλόγου. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ πέρα η κυρία Τεστόρη. Είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και εντωμεταξύ βεβαίως ε, προκύπτουν νέες ειδήσει για, το, για την έκταση του φαινομένου της ε, λάθος σήμανσης. Στο παρελθόν βεβαίως ε, είχαμε σχετική νομοθεσία, σήμανση των τροφίμων. Η συζήτηση τότε βεβαίως αφορούσε το... Πώς θα έπρεπε να σημαίνεται το κρέας, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα είχαν μια θέση διαφορετική από το Κοινοβούλιο. Χτες είχαμε ε, τον τριμερή διάλογο για την σήμανση των βοηδών και το, τα ζητήματα ήταν δύο. Οι κυρώσεις και η χνηλασιμότητα. Γιατί χωρίς κυρώσεις, ε, γιατί αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι πολύ μικρές κυρώσεις, δεν υπάρχει και αποτροπή γιατί είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα. Οι καταναλωτές θέλουν φτηνά τρόφιμα και μετά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σήμερα το πρωί έμαθα πως στη χώρα μου, τη Γερμανία, θα αλλάξει ο νόμος και στο μέλλον όλες οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τον νόμο περί σήμανσης θα κατονομάζονται. Πολύ θετικό αυτό. Όσοι βάζουν ε, και θέτουν σε εμπορία ε, εσκεμένα τέτοια ε, τρόφιμα θα τους αφαιρείται και η άδεια για, να μην τολμάει πλέον κανείς να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Επίτροπο για 10 λεπτά. Μετά θα σας πω ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο και θα δούμε πώς θα μοιράσουμε τον χρόνο μιλίας. Έχουμε μέχρι τις 10.30 γιατί πρέπει να φύγει ακριβώς 10.30 ο κύριος Επίτροπος. Σας έχουμε ακούσει πολλές φορές βέβαια εδώ πέρα στην Επιτροπή μας και χαιρόμαστε για το ότι έρχεστε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να μιλήσουμε. Λοιπόν, ναι, θα σπαταλήσω άλλο χρόνο. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτό το επίκαιρο και ευαίσθητο θέμα, έχοντας βεβαίως πάντα τα πράγματα α, ε, κατά νου όπως είναι στις πραγματικές τους αναλογίες. Έχουμε από τα καλύτερα συστήματα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τις τελευταίες δέκα μέρες μίλησα και στις Επιτροπές Γεωργίας και Γεωργικής Ανάπτυξης ε, και θα ήθελα και σήμερα να ξεκινήσω με τον ίδιο τρόπο. Από τα στοιχεία δηλαδή που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι σήμερα, σχέση με αυτό το σκάνδαλο, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας ή ασφάλειας τροφίμων. Απλά είναι θέμα απάτης ως προς την σήμανση. Δεν είναι θέμα ασφαλής. Γιατί ξέρετε πως το ε, κρέας ε, του αλόγου μπορεί να φαγωθεί και να μπει στο κύμα αρκεί να δηλώνεται στον, ε, στην ετικέτα. Όσοι τρώνε κρέας έχουν το δικαίωμα να ξέρουν αν είναι βόιο, χοιρινό ή αλογίσιο. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που ελέγχουν τα τρόφιμα και τις διαδικασίες οπωσδήποτε φέρουν την κύρια ευθύνη για να ε, διασφαλίσουν το ότι τηρείται ο νόμος. Αλλά Εγώ ρώτησα ποια χώρα είναι υπεύθυνη, αλλά τα λαζάνια αυτά πέρασαν από τέσσερις χώρες και δεν ε, κατονομάσαμε καμία γιατί όλοι κοίταγαν προς μία κατεύθυνση μετά προς την άλλη κατεύθυνση. Οπότε δεν ανέφερα εγώ χώρες και είπα οποιαδήποτε χώρα από την οποία πέρασε αυτό το προϊόν και οποιαδήποτε εταιρεία ε, νεπλάκι ναι, στην παραγωγή, διανομή, αποθήκευση αυτού του προϊόντος ε, είναι ύποπτη. Και ευτυχώς που το είπα γιατί μετά προέκυψε πως έπρεπε να στραφεί σε άλλη ε, κατεύθυνση η έρευνα και τα κράτη-μέλη τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθημερινή εφαρμογή των ε, κανόνων ακριβώς φέρνουν το βάρος ε, αυτό και είναι ευθύνη των κρατών μελών άρα να ελέγξουν αν ένα προϊόν είναι επικίνδυνο και αν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Και είναι γεγονός πως η Κομισιόν έχει την υπηρεσία το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής το οποίο δεν κάνει επιθεωρήσεις, αλλά ελέγχει τους επιθεωρητές στα κρατημέλη, κυρίως για ζητήματα διατροφικής ασφάλειας ε, ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν είναι να κάνουμε εισαγωγή βοδινού από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή, πάνε από την Ιρλανδία στα σφαγεία της ε, Βραζιλίας, της Αργεντινής και τα και ή τα σφαγεία που θα μπορούν να κάνουν την εξαγωγή. Και μετά υπάρχει και το σύστημα γρήγορη ειδοποίηση ε, για τροφές και ζωοτροφές που λειτουργεί αρκετά καλά γιατί παρά το ότι περιορίζεται τυπικά σε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας ε, μόλις προέκυψε αυτό το ζήτημα αυτομάτως ε, για λόγους γνωστοποίησης μεταδόθηκαν τα στοιχεία σε όλα τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν προσεχώς θα παρουσιάσει μία έκθεση για τους ελέγχους που οργάνωσε το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής από πλευράς υγιεινής κυρίως. Όλα τα ευρήματα λοιπόν στην υπόθεση αυτή μεταδοσκαν αμέσω μέσω του συστήματος ΡΑΣ και η Ευρωπόλ συντονίζει την έρευνα για την απάτη και όλα τα κράτη-μέλη θα ενημερώνουν την Ευρωπόλ. Να σας πω τώρα τι συνέβη. Πρώτα απ' όλα είχαμε το περιστατικό της Ιρλανδίας, μετά ακολούθησε 8 Φεβρουαρίου το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 8 Φεβρουαρίου, 13 Φεβρουαρίου Ιρλανδική Προεδρία με τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν έκανε μια έκτακτη, μια έκτακτη συνεδρίαση με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονταν από το σκάνδαλο. Μετά η Κομισιόν πρότεινε στη μόνιμη Επιτροπή Διατροφικής Αλυσίδας μια σειρά επιθεωρήσεων ε, που ξεκίνησαν ήδη και θα κρατήσουν 30 μέρες με την δυνατότητα επέκτασης σε δύο περαιτέρω μήνες. Αυτό έγινε στις 15. 19 του μηνός υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση και υιοθετήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Οπότε ήταν άμεση η αντίδραση. Η Κομισιόν έχει κινητοποιηθεί λοιπόν σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Να εξηγήσω λίγο το εντατικό σχέδιο παρακολούθησης που ξεκίνησε αμέσως. Υπάρχουν δύο σειρές δοκιμών και τεστ σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα τεστ DNA στα βόρεια προϊόντα για να ελέγξουμε το εάν υπάρχει κρέας αλόγου. Θα γίνουν χιλιάδες επιθεωρήσεις, αναλόγως βεβαίως και με τον πληθυσμό των κρατών μελών, τον αριθμό των σφαγίων. Ε, επί τη ευκαιρία να σας πω πως σε όλα τα κράτη-μέλη πλήν της Εστονίας παράγεται αλογίσιο κρέας και βέβαια στο εξάγωνο ή το καταναλώνουν. Και ο απεύθερος έλεγχος αφορά την απουσία φένιλοβοταζόλης ε, στο κρέας, στα σφαγεία ή στα σύνορα. Να σου πω λίγο, ε, γύρω στο 70% του αλλογήσιου κρέατος ε, που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα 30% εισάγεται κυρίως από τη Βραζιλία, Αργεντινή και Καναδά και Μεξικό μικρότερες ποσότητες. Τα τεστ αυτά θα συνεχιστούν για μια περίοδο ενός μηνός με τη δυνατότητα επέκτασης για άλλους δύο μήνες και τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε μέχρι τις 15 Απριλίου και δεσμεύτηκα να τα δημοσιεύσω αμέσως. Δεν έχει νόημα να οργανώνουμε, να πληρώνουμε επιθεωρήσεις και να κρύβουμε τα αποτελέσματα από την κοινή γνώμη. Γιατί θεωρώ πως μόνο η πλήρης διαφάνεια θα ε, αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Όπως είπα θα είναι αναλογικός με το φαινόμενο ο αριθμός των ε, τεστ και όλα αυτά τα υποστήριξαν και τα κράτη-μέλη. Για τα φινιλοβουταζόλη. Συνίσταται να παίρνουμε ένα δείγμα ανά 50 τόνους ε, αλογίσιου κρέατος ε, που έχουν σφαχθεί ή εισαχθεί και ένα ελάχιστο αριθμό 5 τεστ ανά κράτος μέλος. Όταν προκύπτει λοιπόν κύριε Πρόεδρε ένα τέτοιο σκάνδαλο, κάποιοι σπέβδουν να συμπεράνουν πως φταίει το νομοθετικό σύστημα και το νομοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή όμως η ίχνηλασιμότητα ήταν άμεση. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο να βρούμε το από πού ξεκίνησε και Στη συνέχεια έτυχε επεξεργασίας και μετά αποθηκεύτηκε το προϊόν. Οπότε υπάρχει νομοθεσία, το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η απάτη προκύπτει όταν κάποιος ε, παραβιάζει σκεμμένα τους κανόνες. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις ποινικέ κυρώσεις και τη σημασία των ποινικών κυρώσεων. Αν δεν υπήρχε νόμους δεν θα υπήρχαν και κυρώσεις, αλλά ε, βεβαίω η ύπαρξη της απάτης δεν αμφισβητεί την αξία των κανόνων. Και ούτε επίσης πρέπει να υπονομεύει την εσωτερική αγορά. Έχουμε τον πυλόν αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία διακίνησης όχι μόνο ατόμων αλλά και αγαθών και υπηρεσιών και δεν πρέπει να την μονοπεύσουμε. Βεβαίω, μια εσωτερική αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, όταν κάποιο παραβιάζει την νομοθεσία, οι συνέπειε απλώνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στη χώρα όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Και παραλαμβάνω πως έχουμε αναπτύξει από τις καλύτερες νομοθεσίε παγκοσμίω όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα και φαίνεται ότι λειτουργεί το σύστημα από το ότι βρήκαμε αμέσως αυτούς που είχαν εμπλακεί στην αλυσίδα παραγωγής. Με ρώτησαν εάν μου προξένεσε εντύπωση το ότι το ζήτημα αυτό το ανακάλυψαν οι αρχές ενός κράτους μέλους. Είπα δεν με εκπλήσει καθόλου. Είναι ευθύνη των αρχών που ασχολούνται με τη διατροφική ασφάλεια να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία. Και η περίπτωση αυτή ανακαλύφθηκε γιατί σε τυχαίο έλεγχο οι Ιρλανδικές αρχές πήραν τα φτηνότερα βυθέκια που υπήρχαν σε ένα σούπερ μάρκετ και ανακάλυψαν τι συμβαίνει. Όσοι λοιπόν θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν έχει στρατό επιθεωρητών ε, για να εφαρμόζει νομοθεσία είτε σε αυτόν τομέα είτε σε άλλον τομέα πρέπει να ξέρουν πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο για τη διατροφική ασφάλεια, αλλά για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Η ευθύνη παραμένει και πρέπει να παραμείνει στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως η Κομισιόν δεν έχει κανένα ρόλο στον συντονισμό των επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα πριν ή μετά από μια κρίση. Άρα δεν εννοώ και δεν υπονοώ κατά κανένα τρόπο πως ε, πρέπει να χαλαρώσουμε, να ευσυχάσουμε ή πως δεν μπορούμε να αντλήσουμε κάποια διδάγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου τις διαστάσεις των πραγμάτων, να αντιδράσουμε αναλογικά και όχι σπασμωδικά. Ξέρετε, ακόμα σε περιπτώσεις και τέτοιες ακόμα και όταν δεν υπάρχει ζήτημα διατροφικής ασφάλειας, ε, οι αντιδράσεις είναι παράλογες. Και έχουμε και οικονομικές συνέπειες παρά το ότι δεν είναι ζήτημα διατροφικής ασφάλειας. Στο παρελθόν είχαμε ζητήματα διατροφικής ασφάλειας που ο κόσμος ε, αρρώστησε, έχασε τα όργανα του. Ε, εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα, ε, απλά είναι σε μια σοβαρή απάτη ως προς τη σήμανση, γιατί η εμπιστοσύνη του κοινού έχει πληγεί. Και μέρος της διαβεβαίωσης που δίνουμε βρίσκεται ακριβώς στην αντίδρασή μας. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι γρήγορη χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και αναλύοντας τα δεδομένα αμέσως. Καθώς εξελίσσεται λοιπόν το σκάνδαλο, επιβεβαιώνει τη σημασία των σωστών ελέγχων και των αποτρεπτικών κυρώσεων. Ξέρετε πως ε, όταν νομοθετούμε, όταν νομοθετείτε εσείς με μια οδηγία, η οδηγία δεν ε, καθορίζει την φύση των ποινών. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μέλων, αλλά ορίζουμε πως οι ποινές πρέπει να είναι αναλογικές και αποτρεπτικές. Νομίζω η μόνη περίπτωση στην οποία περιγράφηκαν ακριβώς οι ποινές ήταν στην περίπτωση του περιβαλλοντικού δικαίου και εκεί ήταν κανονισμός, όχι οδηγία. Οπότε επαφέτησα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις ε, κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι κατάλληλες και αποτρεπτικές. Και για να ενισχυθεί αυτό η πρόταση της Κομισιόν η οποία θα έρθει για την ενίσχυση των επισήμων ελέγχων θα απαιτήσει από τα κράτη-μέλη να ορίσουν χρηματικά πρόστιμα που θα ε, ισχύουν ε, για την ε, παραβίαση των κανόνων της διατροφικής ασφαλείας στο επίπεδο το οποίο θα αντισταθμίζει την οικονομική ζημία. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο κατάλληλες και αποτρεπτικές αλλά πρέπει να καλύπτουν οι ποινές το όφελος που θα είχε κανείς από την απάτη. Δηλαδή οποιοδήποτε όφελος είχε κανείς από την απάτη πρέπει να ε, αντιστοιχεί στην ε, κύρωση η οποία θα επιβληθεί. Δηλαδή μόνο η προοπτική του να χάσει κανείς περισσότερα από όσα θα κερδίσει από την παρανομία μπορούν να τον αποτρέψουν από το να παρανομήσει. Κάποιοι ζήτησαν περισσότερους επίσημους ελέγχους σε όλη τη διατροφική αλυσίδα. Και εδώ πέρα θα υπάρξουν βελτιώσεις από την ε, επανεξέταση των κανόνων των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή και το σχέδιο παρακολούθησης που πρότεινε η Κομισιόν και δέχτηκαν τα κράτη-μέλη, τι είναι, είναι μια σύσταση της Κομισιόν. Αυτό μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Βεβαίω με σοβαρέ ε, κυρώσει τη τι ε, τωρινέ συνθήκε. Στην πρόταση λοιπόν σκοπεύουμε να δώσουμε Αρμοδιότητε για συγκεκριμένους μόνιμους ελέγχου στην περίπτωση υπάρχει ένας νέος κίνδυνο λαμβάνοντα υπόψη τα τρόφιμα και τις διαδικασίες. Άλλοι ζήτησαν υποχρεωτική σήμανση για την χώρα προέλευσης του κρέατος που περιέχεται σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτό ισχύει σήμερα μόνο για το φρέσκο βόλιο κρέας και θα επεκταθεί τους επόμενους μήνες σε εγωπρόβιο και χοιρινό και προέκυψε η ιδέα η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης να ισχύει και για τα κατεργασμένα προϊόντα, είτε είναι κοιμάς, είτε οτιδήποτε άλλο. Ε, να πω το εξή. Εγώ είμαι ανοιχτό ως προς αυτό το θέμα. Αναμένουμε την αξιολόγηση αντικτύπου. την η οποία βεβαίω απαιτεί νομική προϋπόθεση. Είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες ε, πριν από την υπόθεση αυτή και αναμένουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού την αξιολόγηση αυτή. Αλλά ε, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν σχετίζεται αυτό, όπως σας είπα, με το τρέχον ζήτημα. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε την ε, σήμανση για την προέλευση. Και βεβαίως υπάρχει και η επιπλέον περιπλοκή του τι θα γράφουμε πάνω, πού γεννήθηκε το ζώο, πού το έσφαξαν ή πού έγινε η επεξεργασία. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα δεν αφορούσε την προέλευση, αλλά το είδος του ζώου, του κοιμά. Οπότε, ε, όπως σας είπα, εγώ είμαι ανοιχτός όλες τις προτάσεις και πολλά κράτη-μέλη είναι υπέρ μετά την ε, Συμβουλή Γεωργίας, πρέπει να σας πω, υπέρ της υποχρεωτικής σήμανσης για τη χώρα σήμανσης, αρκεί να εξεταστεί το κόστος, ε, η σκοπιμότητα και ο αντίκτυπος στην εσωτερική αγορά. του υπήν, κύριε Πρόεδρε. Και να με συγχωρείτε. Και όλας γιατί καθυστέρησα. Η εμπιστοσύνη της ε, κοινή γνώμης είναι ένα ευπαθές προϊόν, αν θέλετε, που εύκολα πλήττεται. Ζήτησα από τα κράτη-μέλη να εντείνουν τους ελέγχους τους ε, και να διαχέρουν αμέσως τις νέες ε, πληροφορίες. Φαίνεται λοιπόν πως ε, από τους ελέγχους προέκυψε πως είχαμε λανθασμένη σήμανση 1% βεβαίως και το 1% είναι πολύ αλλά είναι 1% οπότε θα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία των συντομότερων δυνατών για να καθισχάσουμε και τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τους εμπορικούς εταίρους μας. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά το πόσο μεγάλη σημασία έχει να αποκατασταθεί η πλήρης εμπιστοσύνη στη διατροφική αλυσίδα και βασίζομαι στη συνεργασία των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Οπωσδήποτε δεν έχουμε σκάνδαλο τροφίμων αλλά ένα σκάνδαλο απώλειας εμπιστοσύνης δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα οικονομικά. Εγώ αναμένω τα νούμερα και από τους γεωργούς ε, και τις εκμεταλλεύσεις το τι δηλαδή μείωση του τζίρου θα έχουμε. Θα είναι μεγάλη ζημιά. Εντάξει στιγμής βεβαίως είναι καθυσυχαστικά τα νούμερα αλλά φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη δυσπιστία το έζησα και στο δικό μου το κρατήδιο. Ε, αυγά είχαμε με λάθος σήμανση. Οπότε νομίζω πως απαιτείται να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Και νομίζω πως και ο κλάδος πρέπει να ε, δείξει την ε, ετοιμότητα να διορθώσει τα πράγματα γιατί βλέπουμε πως καμιά φορά ξέρεις, ξέρετε είχαμε σκάνδαλα μόλιβδο σε αυγά ειδικά στον τομέα των ε, έτοιμων ε, και επεξεργασμένων ε, τροφίμων θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η ίχνη και να μπορεί να αποδεικνύει κανείς ότι τι υπάρχει μέσω στο προϊόν. Ε, οπότε δεν υπάρχει, όπως είπαμε, πρόβλημα υγιεινής ε, των τροφίμων, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνη. Και πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ε, με την εχνηλασιμότητα να γνωρίζουμε το τι γίνεται, πού, στη διατροφική αλυσίδα, αλλά και με κυρώσεις. Στις κυρώσεις πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, με περισσότερο αποτρεπτικό χαρακτήρα. Είδατε πού πήγε ε, ε, το, το κρέας ε, ζαλίζεται κανείς με το να παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδρομή. Τέλος πάντων, δεν θα βγάλω κι εγώ τη δική μου ομιλία, θα διαβάσω τώρα τα ονόματα που είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Εάν κάποιος δεν άκουσε το όνομά του, παρακαλώ να το πει. Λίνα Μεκέμπεν, Λίνα Μακάβαν, Κορίν Αννα και Χίτα Αλεσούζα για την Γκουε. Αυτοί είναι οι συντονιστέ. Και μετά. Μετά, περιμένετε. Πίλα Αιούζο, dann Marek Demes Mecker, dann Christel Schaldemose, dann die Kollegin McGuinness, Paulsen, Okoni, Hibner, Nicholson, Würmert, Pagnot, Sofolokleos, dann Pock, Lepage hatten wir schon, Toni Manders und dann Frederik Ries. Η πώς μπόρεσα να την ξεχάσω. Και Μαριέτα Ουλσκούκ. Ξέχασα κάποιον. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές. Δύο λεπτά. Λίντα Μακάβαν. auch mit Γιατί έχει και το άλλο θέμα Ευχαριστώ. Κύριε Πετροβά. Στην Κλένης Γκούλμαν θα αφήσω το θέμα της επισήμανσης ε, ε, των τροφίμων, γιατί είναι συγκέντρια των σοσιαλιστών για το θέμα αυτό και σίγουρα διαφωνεί με, με πολλά σημαντικά θέματα που είπατε. Και θα μιλήσει αργότερα η κυρία Γουίλμον, ότι είναι στον κατάλογο. Είπατε ότι βρέθηκε το πρόβλημα με κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους στην Ιρλανδία. Και μετά μας είπατε ότι όλο το σύστημα της επιστημιστικής ασφάλειας είναι το καλύτερο στον κόσμο και ότι δεν χρειάζεται και πολλές αλλαγές αυτό. Διαρωτώ με όμως. Γνωρίζουμε πόσοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο συστηματική είναι αυτή η τυχαία έλεγχη. Πόσα κράτη-μέλη πραγματοποιούν τέτοιου τυχαίου ελέγχου, κρατούν ε, στοιχεία και αρχεία, γιατί ξέρω ότι μερικέ ε, χώρε περιορίζουν αυτού του δειγματοληπτικού ελέγχου. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για πόσο καιρό έγινε εσφαλμένη επισήμανση ε, του κρέατος αυτού. Και τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, πώς είναι σίγουρο θα αποτρέψουμε επανάληψη ε, της κατάχρησης αυτής αν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου. Προσπαθείτε να περάσετε την ιδέα ότι το σύστημα είναι σωστό, αλλά δεν νομίζω ότι συμφωνούν μαζί σας οι καταναλωτές. Δεν νομίζω ότι πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι το σύστημά μας ε, για την ιχνηλασιμότητα μέχρι το σφαγείο είναι άψογο. Και μας είπατε ότι βρέθηκε βέβαια το κρέας, αλλά ούτως ή άλλως ε, ο κοιμάς είναι ένα μεταποιημένο προϊόν που έχει κυκλοφορήσει παντού και τελικά χάνουμε την χρυλασιμότητα. Δεν ξέρουμε από πού πραγματικά ξεκίνησε. Πραγματικά πιστεύετε δεν έχουμε πρόβλημα στην επιστηστική μας αλυσίδα. Τζέβερ, ευχαριστώ τον κύριο Πίτροπο που ήρθε, αλλά οτι δεν εχουμε προβλημα στην επιστηστικη μας αλυσιδα ευχαριστω τον κυριο πιτροπο που ηρθε αλλα δεν ξερω αν μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας των τροφίων και είναι μόνο ζήτημα σήμανσης πρέπει να δούμε το ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και υπάρχει και οικονομική ζημία ήδη. Άρα είναι ένα διατροφικό σκάνδαλο. Και δεν ξέρω αν το συμπέρασμα είναι ε, ήταν μια εγκληματική ενέργεια και αυτό δεν μπορεί να το εμποδίσει κανείς με τους νόμους, είναι εξορισμό παράνομο. Νομίζω πως ένα συμπέρασμα είναι πως ε, θα πρέπει να δούμε την αλυσίδα του ελέγχου αυτού ε, που πρέπει βεβαίως να καθορίζεται από την Ευρώπη και να την εκτελούν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το πόσο συχνά και το πώς πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι πρέπει να το ορίζει ο Ευρωπαίος νομοθέτης και γνωρίζουμε και από άλλους ε, τομείς πως δεν μπορούμε να ελέγχουμε 100% αλλά θα πρέπει όπως είπα να φτάσουμε το σημείο εκείνο στο οποίο η παρανομία θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα πρέπει να βρεθεί δηλαδή μαθηματικά ο τρόπος. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία συνολικά να επανεξετάσουμε την σήμανση των ε, τροφίμων και οπωσδήποτε αυτός είναι ένας παράγοντας που θα εμποδίσει να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι βιομηχανοποιημένη η παραγωγή των τροφίμων και πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό α, μπορούν να δεχτούν κάτι τέτοιο οι καταναλωτές. Και νομίζω πως ο καταναλωτής έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Μακροπρόθεσμα δηλαδή για να επηρεάσει τις ε, συμπεριφορές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ήρεμη ανάλυση και βεβαίω όπως είπατε και εσείς δεν είχαμε κάποια βλάβη στην ανθρώπινη υγεία οπότε μπορούμε να μας στοιχειώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ να πάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Μας είπατε ότι θεωρείτε ότι η νομοθεσία μας είναι καταπληκτική. Δεν με πείσατε. Γιατί αν ε, ευσταθούσαν αυτά που λέγατε θα τα πίστευαν και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Σίγουρα νομοθεσία έχουμε, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί. Η κυρία Βιλμότ θα μας μιλήσει για το θέμα της επισήμανσης των τροφίμων. Ακόμη κι αν έχουμε την καλύτερη νομοθεσία του κόσμου, από τη στιγμή που δεν ασκείται έλεγχο, είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Ω εκ τούτου είναι εύκολο και συμφωνώ με τον προλαλήσαντα να θεωρούμε ότι πρόκειται για απλή απάτη και από τη στιγμή που υπάρχουν απαταιώρες στον κόσμο τι να κάνουμε. Συγγνώμη κύριε Επίτροπε, αλλά δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Όταν διαβάζουμε το διεθνή τύπο στα τέλη του 2010, το γαλλικό, τον αγγλικό τύπο, ακόμη και τον αμερικανικό, Βλέπουμε την περίπτωση των, των ελλαδικών αλόγων και το, της φαγής τους που επεκτάθηκε παντού, εξαπλώθηκε παντού. Και γνωρίζετε και η Επιτροπή γνώριζε ότι είχαμε ουσιαστικά δεκαπλασιάσει τη σφαγή αυτών των αλόγων. Πού πήγαν αυτά τα άλογα, διαρωτηθήκαμε τότε πώς διοχετεύθηκε αυτό το, ή πού διοχετεύθηκε αυτό το κρέας. Μήπως διοχετεύτηκε στην επισητιστική αλυσίδα. Προβληματιστήκαμε τότε όπως θα έπρεπε αν ε, ζώα που δεν προορίζονται για σφαγή και άρα δεν ε, ε, έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτά που προορίζονται για σφαγή, παρόλα αυτά καταλήγουν στην επιστηστική αλυσίδα, όπως η περίπτωση της φαινιλομπουταζόλης δεν νομίζω ότι εξετάσαμε τι έγινε, ούτε το διερευνήσαμε. Οπότε ανακύπτει το θέμα του ελέγχου. Είναι πανεύκολο να νομοθετούμε και να παραπέμπουμε στα κράτη-μέλη το θέμα της εφαρμογής και του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Γνωρίζουμε, εκτός και αν θέλουμε να θελοτυφλούμε, ότι με τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας αναγκάζονται να, περιορίσουν τον αριθμό των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με, την, με τις επιθεωρήσεις, του ελέγχους και τις επαληθεύσεις. Οπότε ουσιαστικά η νομοθεσία μας παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι εικονική, ενώ αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι μια έμπρακτη εφαρμογή της νομοθεσίας μας. Έχω λοιπόν δύο-τρεις ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναθεωρήσει το κείμενο για την ενημέρωση του καταναλωτή. Πώς θα ελέγξετε την εφαρμογή της νομοθεσίας, ε, θα εξακριβώσετε την εφαρμογή της από τα κρατημέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βιβλιάριο υγείας των ζώων που προορίζονται για σφαγή. Είναι ε, συμβατά με την νομοθεσία αυτά τα βιβλιάρια υγείας. Πώς θα αποφύγουμε μετάδοση προβληματικού κρέατος στην επιστημιστική έλυση. Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας. Και με αγριοκοιτάει η κυρία Γκροστέτ. Δεν θέλω να ρισκάρω το κάτι τέτοιο πρωί-πρωί. Αρτ Στάς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι νομίζω ένα διατροφικό σκάνδαλο, το σκάνδαλο αυγών, βοδινού κτλ. Έχετε κάποια εικόνα, όπως είπε και η κυρία Μακάβαν, για τις επιθεωρήσεις των ε, κρατών μελών, γιατί όλα τα κράτη-μέλη κάνουν οικονομίες. Πόσοι επιθεωρητές υπάρχουν, πόσες επιθεωρήσεις γίνονται, αυξάνονται οι έλεγχοι, μειώνονται οι έλεγχοι, υπάρχουν καλά κράτη-μέλη, κακά κράτη-μέλη ως προς επιδόσεις τους. Δεύτερον, έχουμε τους ελεγκτές των ελεγκτών, την υπηρεσία αυτή στην Ιρλανδία, αλλά και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κόβουμε. Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε πως ε, δεν θα υπάρξει περικοπή στο ε, Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικής όσον αφορά τα κονδύλια και το προσωπικό. Μετά, τι γίνεται με τις συστάσεις που κάνει το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικής κάνει 300 επιθεωρήσεις το χρόνο. Δίνεται συνέχεια. Μήπως να πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός έλεγχος, να κάνουμε εμείς ε, κάθε χρόνο μια συζήτηση στην Επιτροπή μας για το πώς λειτουργεί το Γραφείο Τροφίμων και Εκτινιατρικής για να ξέρουμε τι γίνεται. Επίσης λέτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μέχρι σήμερα ναι, αλλά πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απαταιώνες που το έκαναν. Έτσι, γιατί να σεβαστούν και τους κανόνες της υγιεινής, ε, για τις ορμόνες ε, και λοιπούς ε, παράγοντες ε, αυξητικούς. Επίσης, μην ξεχνάμε πως ε, μεγάλο τμήμα του αλογίσιου κρέατος που καταναλώνεται εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν ε, άσχημε εκθέσει από το Γραφείο Τροφιμών και Κτηνιατρικής για τι εισαγωγέ από Καναδά και Μεξικό. Πώς σίγουροι είμαστε. Ευχαριστώ, Άννα Ροσμπαχ. Er- Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι συμφωνώ πλήρω με τον Πρόεδρο που μίλησε για έλλειψη, ανάγκη, έλλειψη εμπιστοσύνης, για δυσπιστία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας μιλήσατε για τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας κάνατε μια γενική επισκόπηση για το θέμα, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι είστε ανοιχτό στο θέμα της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών. Αλλά πιστεύω ότι ε, όταν αγοράζουμε λουκάνικα θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς, από, τι ακριβώς αποτελούνται. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ε, αναφέρει η ετικέτα τη σύσταση του προϊόντος. Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι αγοράζει και τι τρώει. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε και εισαγόμενα προϊόντα και τι ακριβώς αναφέρει η ετικέτα, γιατί η ετικέτα δεν αναφέρεται μόνο στη χώρα προέλευσης. Στο μεταξύ έχει περάσει το προϊόν και μπορεί να συνεχίζει τη μεταπίση του και από αλλού. Ποιος θα ασκεί τον έλεγχο, θα πρέπει να βρούμε μια συνολική λύση. Όπως είπατε, έχουμε τους μηχανισμούς και τη σωστή νομοθεσία. Πώς όμως θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της, πώς θα μεριμνήσουμε ώστε όλα τα κρατη την εφαρμόζουν σωστά και πώς θα βεβαιωθούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με την κοινωτική νομοθεσία για τους προδιαγραφές σφαγής και της ετικετοθεσίας. Ευχαριστώ. Εξοικονομήσατε τα 20 δευτερόλεπτα της Κόριν ε, Λεπάζ, οπότε ακολουθεί η επόμενη συνάδελφος. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις στον Επίτροπο. Πρώτον, μας είπατε κύριε Επίτροπε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία είναι αρκετή και ότι το μόνο που θα πρέπει να προσθέσουμε είναι η υποχρεωτική αναφορά της χώρας προέλευσης στην ετικέτα. Μήπως ήταν πολύ πιο λογικό, πολύ πιο συνετό και πολύ πιο χρήσιμο για τη δημόσια υγεία να έχουμε ένα κεντρικό μητρό, ένα κεντρικό αρχείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σε σχέση με τα ε, υγειονομικά βιβλιάρια των ζώων, εν προκειμένου των αλόγων. Γιατί με ένα τέτοιο κεντρικό μητρό θα ήμασταν σίγουροι ότι ζώα που δεν έχουν επιλεγεί για σφαγή, όντως δεν ε, θα διοχετεύονται στην ε, επιστημιστική αλυσίδα, ενώ όσα διοχετεύονται θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές. Δεύτερη ερώτηση. Μας διαβεβαιώσατε ότι το θέμα δεν είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας ή επιστημιστική ασφάλειας. Μου φαίνεται παράδοξο που ισχυρίζετε κάτι τέτοιο. Πώς δικαιολογείτε τότε ότι ο Οργανισμός για την Επιστημιστική Ασφάλεια προειδοποίησε τις γαλλικές αρχές ότι βρέθηκε φενιλό στο αλογίσιο κρέα και ότι παρισέφρεσε στην επιστημιστική αλυσίδα. Μήπως δεν μας λέτε την αλήθεια. Και θα πρέπει αυτό το θέμα οπωσδήποτε να, χρησιμο... να αναφερθεί ως θέμα που έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία. Και ένα σχόλιο. Ο Γερμανός Υπουργός δήλωσε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι ναι μεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά το ύποπτο κρέας που αποσύρεται από την αγορά θα μπορούσε να μοιραστεί στους απόρους. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι στην Ευρώπη έχουμε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και σε περίπτωση της κρίσης θα πρέπει τους φτωχούς, τους απόρους να τους πλήξουμε ακόμη περισσότερο μοιράζοντάς τους μολυσμένο κρέας. Παρακαλώ μη φωνάζετε γιατί είναι δύσκολο και στα ακουστικά. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πίτροπο να απαντήσει στον πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων. So been, have... Ναι, γιατί πάρα πολλά ζητήματα ετέθησαν. Ξεκίνησα την παρέμβασή μου λέγοντας πως έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Και το εννοούσα, όμως δεν θα πρέπει να ε, είμαστε αυτάρεσκοι και να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, γιατί είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση ε, σκανδάλου ή κρίσης. Πάντως, όπως σας είπα, ε, δεν είναι πρόβλημα νομοθεσίας, γιατί υπήρχαν κάποιοι που είπαν και ότι αν είχαμε διαφορετική νομοθεσία δεν θα είχε προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει η νομοθεσία, είναι καλή νομοθεσία, απαιτεί την επισήμαση των ζωικών συστατικών σε κάθε προϊόν. Φυσικά είναι θέμα επιβολής. Αλλά υπάρχουν και όρια στο κατά πόσο μπορεί η επιβολή να εγγυηθεί την πλήρη συμμόρφωση. Έχουμε μια νομοθεσία κατά των κλοπών, αλλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται κλοπές. Δεν σημαίνει πως η επιβολή δεν είναι σωστή ή αποτελεσματική. Και αν θέλατε να με ζητήσετε ε, διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο δεν ξανασυμβεί, μα δεν μπορώ να σας δώσω τέτοια <laughs> διαβεβαίωση. Από τη στιγμή που υπάρχουν εταιρείε, κόσμος έξω που προσπαθεί να παραβιάσει την νομοθεσία. Φυσικά και πρέπει να το κάνουμε πιο δύσκολο, να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν καταλήλως όλοι αυτοί, αλλά όταν ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας ότι δεν είναι θέμα ασφάλειας των τροφίμων μέχρι στιγμής, το είπα, διότι από τις ενδείξεις που έχουμε δεν πρόκειται για θέμα ασφάλειας των τροφίμων. Αντιθέτω, θα πρέπει να πούμε ότι το σύστημά μα λειτουργεί όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό βέβαια θα πρέπει να επισκιάσει το άλλο θέμα τη απάτη, εφόσον αυτή υπήρχε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν θέμα αμέλεια. Ήταν η θελημένη απάτη για ε, μεγαλύτερο κέρδος, γιατί το, το άλογο ε, κοστίζει λιγότερο από το βόδι. Αυτό είναι εις βάρος του καταναλωτή. Θέλησαν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα αυτοί οι κύριοι. Λοιπόν, το δεύτερο, ε, η δεύτερη εντύπωση που είχα με βάση τον τόνο των ερωτήσεών σας είναι περιμένετε τα κράτη-μέλη να τα κάνουν όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε η Κομισιόν να αναμειχθεί περισσότερο. Κοιτάξτε, αν τα κράτη-μέλη δεν έχουν την διοικητική δυνατότητα, ικανότητα να κάνουν αυτό που ο νόμος τους επιβάλλει να κάνουν, δηλαδή να επιβάλλουν την νομοθεσία, Φανταστείτε, ξέρετε τι οικονομικές και ανθρώπινες δυνάμεις έχει η Κομισιόν ώστε να αναμειχθεί άμεσα και να εφαρμόσει άμεσα εκείνη αυτή την νομοθεσία. Εντάξει, άμα σας έλεγαν ναι, θα δω τι θα κάνω, θα σας ξεγελούσα, θα σας δημιουργούσα ε, ε, ε, λάθος φρούδες ελπίδες. Ε, ξέρετε πώς πάει το σύστημα. Η Κομισιόν προτείνει την νομοθεσία, την εγκρίνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και μετά εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Αν τα κράτη-μέλη επανειλημμένως και ηθελημένα αγνοούν την νομοθεσία, ε, τότε η Κομισιόν φροντίζει ώστε να τους πάει στο δικαστήριο. Αλλά η πρώτη γραμμή της επιβολής απαραίτητος εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Εκτός φυσικά αν προκύψει ιδέα όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για κάθε ζήτημα, κάθε είδους νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φτιάξουμε ένα μια τεράστια υπηρεσία επιβολής που θα παρεμβαίνει, θα εκτελεί άμεσα την περιβαλλοντική νομοθεσία, την ε, νομοθεσία περί ασφάλειας των τροφίμων, την νομοθεσία ε, όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν λοιπόν υποκριτικό να σας πω ότι αυτό δεν είναι, ε, ότι αυτό είναι δυνατόν. Δεν γίνεται ούτε για τούτη την περίπτωση, ούτε για οποιαδήποτε περίπτωση κάτι τέτοιο. Δεν θέλω λοιπόν να δημιουργήσω ελπίδες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε περισσότερο τα σχέδια και τα προγράμματα επιθεωρήσεων των κρατών μελών. Επιβάλλονται τυχές επιθεωρήσεις για τα προϊόντα κρέατος και το κρέας που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τέτοια σε εκθέσεις. Ε, Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση του, κατα... του αν έχουμε πληροφορίες για το πόσες επιθεωρήσεις γίνονται ετησίως. Ναι και είναι δημοσιευμένα τα στοιχεία και έχουμε δημοσιεύσει και τα περσινά στοιχεία. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή γίνονται οι επιθεωρήσεις αλλά και υπάρχουν και... Ε, ποινές ε, αποτροπής ε, σε σοβαρές ότι δεν θα ξανασυμβεί. Και για τις κλοπές, όπως σας είπα, υπάρχουν ποινές που προβλέπονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αποτρέπονται όλοι από το να κλέψουν. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε ότι οι ποινές θα εφαρμόζονται. Αντίθετα με το τι γίνεται σε χώρες τώρα εκτός της Ένωσης, οι τυχές επιθεωρήσεις δεν γίνονται στο τέλος της αλυσίδας ε, ε, τροφίμων, αλλά σε κάθε φάση και σε κάθε μια φάση έχουμε συγκεκριμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις. Έπειτα το θέμα είναι αν παρακολουθούνται η κίνηση των αλόγων και αν υπάρχει εχνηλασιμότητα. Ναι, υπάρχει σύστημα το οποίο απαιτεί διαβατήριο για το κάθε άλογο και εκεί συμπεριλαμβάνεται η πληροφόρηση για το τι τρώνε τα άλογα, πώς τρέφονται αυτά τα άλογα. Είναι υποχρεωμένα τα κρατημέλη να καταγράφουν ε, την διατροφή τους και έτσι και ξέρουμε αν συγκεκριμένα φάρμακα έχουν μπει στο σύστημα σε αυτή την περίπτωση ας πούμε αν έχουν πάρει συγκεκριμένα φάρμακα τα συγκεκριμένα άλογα και υπάρχουν και κανόνες επί όλων αυτών. Για ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην τελευταία λήψη του συγκεκριμένου φαρμάκου και του σφαγίου και σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να μπει αλογίσιο κρέας στη δροφική αλυσίδα αν έχει χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Αποκλείονται πλήρως δηλαδή ορισμένα φάρμακα από την ε, διατροφική αλυσίδα. Υπήρξε και μια ερώτηση για το μέρος προέλευσης. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να προτείνω τέτοια νομοθεσία. Πρέπει αυτό να είναι σαφέ. Το μόνο που λέω, και έχω και ανοιχτό μυαλό για όλα αυτά, για όσου είπαν ότι είμαι ότι κολυσιεργό κτλ. Δεν αληθεύει. Αντιθέτω, ε, θα προσπαθήσουμε να δούμε την έκθεση για την ε, αντίκτυπο πριν από την προθεσμία. Και η νομοθεσία αυτή ισχύει εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια πριν συμβεί κάτι. Και δεν είναι κάτι νέο, είναι ένα παλιό θέμα, το οποίο βέβαια τώρα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία λόγω αυτής της κρίσης. Αυτό που τόνισα στις δημόσιες μου δηλώσεις είναι ότι δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση πως αυτό το περιστατικό συνέβη επειδή δεν υπήρχε νομοθεσία για την ε, επισήμαση του ε, ε, μέρους προέλευσης του ζώου σε αυτά τα προϊόντα που περιέχουν κρέα. Γιατί θα ήταν άδικο να κάνουμε τέτοιο. Αν θέλετε να μεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για οποιοδήποτε λόγο για να πετύσετε επιτάχυνση τη νομοθεσία για την επισήμαση ώστε να συμπεριληφθεί και το μέρο προέλευση, εντάξει. Γιατί όχι, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Μην περιμένετε ότι θα είναι εύκολο. Υπάρχουν θέματα που αφορούν εσωτερική αγορά, το κόστος του συστήματος, ποιος θα, το, θα επιβαρεθεί με αυτό δεν θα είναι εύκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε. Έχω ήδη ενημερώσει την Επιτροπή σα ότι αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών, όχι όλα, αλλά και μάλιστα ορισμένα έχουν αλλάξει και τη θέση του, την προηγούμενη, είναι υπέρ Πάντως δεν είναι η αρχή, ούτε είναι το αίτιο αυτό το περιστατικό και υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν. <laughs> Ναι. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν πού που, από πού προέρχεται αυτό το ε, κρέας. Από το Μάλτα, από την οποιαδήποτε χώρα αυτό πρέπει να συζητηθεί και ε, όπως σας είπα έχω είμαι απόλυτα ανοιχτός. Απλώς ήθελα να δηλώσω πως δεν θα είναι εύκολη η υπόθεση. Δεν είναι εύκολο, είναι περίπλοκο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτή την έκθεση τον Μάιο τον Ιούνιο όπως θα περιμέναν κάποιοι αλλά όσο γίνεται πιο σύντομα. Για την τελευταία ερώτηση που άκουσα για το τι είπε ο Υπουργός, Γερμανός Υπουργός Ανάπτυξης για το τι θα κάνουμε με το κρέας το οποίο αποσύρθηκε από τις αγορές αλλά που είναι απόλυτα ασφολές για ανθρώπινη κατανάλωση. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι θέμα των κρατών μελών να το αποφασίσουν με την προϋπόθεση ότι τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή, αν πουλάς ή δίνεις δωρεάν αλογίσιο κρέας θα πρέπει να το λες ότι είναι κρέας και όχι άλλο. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Πρέπει να περιοριστεί ο καθένας σε ένα λεπτό στην ερώτησή του για να μιλήσουν όλοι. Ή αλλιώς δεν θα μιλήσουν όλοι και θα μιλήσουν οι μισοί. Άντες Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο να ζει κανείς. Αλλά υπάρχουν εύκολοι τρόποι για να ζει κανείς. Με το καλύτερο σύστημα επιστηστικής ασφάλειας του κόσμου και με το καλύτερο σύστημα επισήμασης είχαμε απάτη που δεν είναι απειρολάγιστη η ε, μικρή ή η μεγαλη Είναι απάτη, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εδώ δεν έλειπε η σήμαση, η ετικέτα, η χώρα προέλευσης. Η έλεγχη ήταν αυτή που δεν ε, ήταν αποτελεσματική. Το θέμα είναι με περισσότερους ελέγχους, με περισσότερες επιθεωρήσεις να ανακαλύπτουμε τις απάτες και όχι να μην, να μην έχει νόημα να το κάνουμε. Γιατί αν δεν καλύψουμε τα κενά θα συνεχιστούν τα φαινόμενα της απάτης. Θα πρέπει να αυξήσουμε τους ελέγχους και να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιούν τη λιτότητα ως άλοθη ή ως προθάλαμο της απάτης. Γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορεί να κάνει συστάσει και παροτρύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι σαφέ ότι το πρόβλημα δεν αφορά την ε, νομοθεσία, ούτε θα επιληθεί με περισσότερη νομοθεσία, ούτε με την επισήμαση της χώρας προέλευσης. Ζητούμε ελάφρυση της γραφειοκρατίας. Δεν μπορούμε να ζητούμε αύξηση της ε, νομοθεσίας. Είναι συνεπές. Άλλωστε, αυτός που ε, πληρεί μία νομοθεσία, πληρεί και τη δεύτερη ή και το αντίθετο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερο συντονισμό των επιθεωρήσεων ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και κρατών μελών. Και επίση να επιβληθούν κυρώσει για να μην έχει συμφέρον ο ανέντιμο εμπορο να πραγματοποιήσει τέτοια παράνομη χροκερδή συμπεριφορά. Υπάρχουν κενά και αδυναμίε. εξού και η κακή διαχείριση του συστήματο έγκυρης προειδοποίηση. Δεν ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, αλλά είχαμε άλλα πρόσφατα παραδείγματα που δημιούργησαν τεράστια οικονομικά προβλήματα και προκαλούν σύγχυση στον καταναλωτή. Και το θέμα αυτό δεν είναι μόνο απάτης, είναι θέμα ασφάλειας της επιστηστικής αλυσίδα. Από πού προήλθαν αυτά τα άλογα, πώς μπήκαν στην επιστηστική αλυσίδα, κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίζει το θέμα και να διαχειρίζεται καλύτερα του, τους κινδύνους. Δεν είναι τα κράτη-μέλη επιφορτισμένα με αυτό. Μάρεκ Ντέμεσμέκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ακριβώς στον έλεγχο και στις κυρώσεις. Και εγώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν και τη διαφάνεια που εξαγγείλεται. Αλλά μην ξεχνάμε ε, πως ε, θα δημιουργηθούν έτσι και διοικητικά βάρη, ειδικά για τις μικρές ε, επιχειρήσεις. Τώρα, για την ε, σήμανση είπατε πως ε, αναμένονται εντό του έτους νέες προτάσεις. Πώς θα φροντίσετε έτσι ώστε ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις να μην επιβαρυνθούν διοικητικά. Και όσον αφορά επίσης την πολυπλοκότητα της διατροφικής αλυσίδας. Ε, ως ε, φλαμανδός βουλευτής εγώ είμαι υπέρ μιας πιο σύντομης και ε, απλούστερης διατροφικής αλυσίδας και έτσι θα ε, είναι τα προβλήματα λιγότερα και θα έχουμε ίσως και έναν ε, και άλλους τομείς να αναπτυχθούν. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι το θέμα είναι πρωταρχικά θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά αν οι καταναλωτές δεν μπορούν ε, να εμπιστευτούν την, ε, την ενιαία αγορά, τότε η ακαιρεότητά της ε, υπονομεύεται. Μπορούμε να εγκρίνουμε ένα σύστημα ώστε να καταδεικνύουμε τους ενόχους, να μπορούν να το ελέγχουν οι καταναλωτές. Και μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο υπόλοιπο τμήμα τη επισήμασης, την αναφορά της περιεκτικότητα σε λίπο, σε άλλες ουσίες, γίνονται σωστοί έλεγχοι σε όλα τα κρατημέλη. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Γιατί αν μπορεί κανείς να κλέψει στο κρέα, μπορεί να κλέψει και σε άλλα συστατικά. Η κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχω πέντε ερωτήσεις, αλλά προτιμώ να σα τη στείλω γραπτό παρά να χάσουμε ώρα εδώ. Νομίζω ότι κάτι που παραλείψαμε είναι το 2004 και θα ήθελα να το σχολιάσει ο Επίτροπος. Ο κανονισμός του 2006 έλεγε ότι όλες οι άδειες σε μεταπητικά εργοστάσια θα ελέγχονται ε, μία φορά το χρόνο και θα γίνεται και προαγγελία ελέγχων. Προηγουμένως είχαμε επιθεώρηση καθημερινή γιατί περί αυτού πρόκειται. Μιλήσατε για δειγματοληπτικού ή τυχαίους ελέγχους. Πολύ καλή φράση αυτή. Τυχαίος έλεγχος, δειγματοληπτικό. Το θέμα τη επιθεώρηση έχει νευραλική σημασία, του ελέγχου. Ποια είναι τα σχόλιά σα για τη συχνότητα. Και κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη μου πρόβλημα υπάρχει στην επισήμανση. Και ίσω σοκάρω μερικού, αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η επισήμανση και όχι η λύση. Και το Συμβούλιο κατέληξε σε κακέ λύσει θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα σας αποστείλω πάντως και γραπτό στι πέντε ερωτήσεις μου για τις οποίες περιμένω και απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το θέμα δεν αφορά το κρέας, αλλά την εμπιστοσύνη του κοινού. Συμφωνώ πράγματι με αυτό. Αλλά ταυτόχρονα Έρχεται εδώ πέρα η Κομισιόν και μας λέει πως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα ή τα ΜΜΕ. Όχι, εγώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Επίτροπος έχουν ευθύνη. Αυτό θέλουν οι, οι καταναλωτές όταν ε, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά ε, τροφίμων. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Να ξέρουμε τι αγοράζουμε. Και να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση σε όλο το κρέας. Είτε είναι ε, φιλέτα, είτε κοιμάς, είτε έτοιμα γεύματα. Γιατί βεβαίως πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στο σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων και χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Πάλσεν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Νομίζω πρέπει να παραδεχτούμε πως ε, τα τρόφιμα δεν είναι ένα απλό προϊόν και οι άνθρωποι δεν είναι μόνο θέμα βιολογίας. Έχουμε μια γενετική κληρονομιά που σημαίνει πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι τρώμε και στο τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Και στη σημερινή κοινωνία ένας ε, απλός άνθρωπος δεν έχει την παραμικρή ελπίδα να γνωρίζει τι βρίσκεται μέσα στη συσκευασία που αγοράζει. Δεν μπορεί να τα μυρίσει το, το φαΐ, δεν μπορεί να το αγγίξει, βασίζεται μόνο στις πληροφορίες που γράφει πάνω η ετικέτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα ασφάλειας, όχι, εντάξει, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης. Και όταν μιλάμε για την σήμανση πρέπει να είμαστε πολύ σκληρότεροι στους ε, ελέγχους ναι να γίνουν στα κράτη-μέλη, αλλά χρειάζεται και επιθεώρηση της εσωτερικής αγοράς διασυνοριακή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που είστε σήμερα εδώ. Εγώ είμαι εισηγήτρια για τον ε, ισχύοντα κανονισμό που σχετίζεται με την επισήμανση του βοήου κρέατος ε, ε, είχαμε τριμερή διάλογο εχθές. Θα πρέπει να σας πω πως είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ακούω, γιατί άκουσα το σύνολο των ομάδων να συμφωνούν σε ένα πράγμα. Ότι το πρόβλημα αφορά τον έλεγχο και την ποινή, την κύρωση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κομισιόν αυτό να το εισακούσει, δηλαδή ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ενίσχυση των ελέγχων και των διοικητικών κυρώσεων που είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν και πρέπει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσουν τα κρατημέλη ώστε να ελέγξουν καλύτερα και να ε, τιμωρήσουν καλύτερα και να έχουν και τη ε, μέσα για να το κάνουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αποκομίσουμε διδάγματα από την επικαιρότητα, να μην κάνουμε ε, κινησιακές κινήσεις, γιατί πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσουμε από την απάτη, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι έτσι. Και ε, σας παρακαλώ κύριε Επίτροπε, ε, ακούστε, ακούστε αυτό που σας λέμε για τους ελέγχους και τις κυρώσεις. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία Χίμπνερ, ευχαριστώ και ε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο που επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για παραβίαση Τη ασφάλεια των τροφίμων, γιατί αυτό πραγματικά θα ήταν έγκλημα ει βάρο των καταναλωτών. Το αλογίσιο κρέα ε, έχει μεγάλη θρεπτική αξία, αλλά εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη απάτη, μια εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, η εσχροκέρδεια είτε παραγωγών είτε των μεταπίτων προκάλεσε αυτό το φαινόμενο της καταχρηστικής ε, χρήσης αυτού του βολογησίου κρέατος. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο και πώς θα συντάξουμε νομοθετικές διατάξεις ώστε να στεγανοποιήσουμε το σύστημα του ελέγχου. Και δεύτερον, με ποιο τρόπο ε, θα θεσπίσουμε και ένα σύστημα κυρώσεων που ε, δεν θα ενθαρρύνει ε, αυτούς που είναι διατεθειμένοι να κάνουν απάτες να αναλάβουν τον κίνδυνο θα πρέπει να είναι υψηλές οι κυρώσεις και βαριά τα οικονομικά πρόστιμα. Κύριος Νίκολσον, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Επίτροπος είχε δίκιο ότι όταν είπε ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα. Όμως οι εγκληματίες, οι απαταιώνες, στην ουσία περνάνε τον καιρό τους προσπαθώντας να παραβιάσουν ακόμα και τα καλύτερα συστήματα. Και ό,τι σύστημα και αν φτιάξουμε, πάλι θα προσπαθήσουν να το παραβιάσουν. Μη, κάνατε ένα σχόλιο για τα διαβατήρια των αλόγων αλλά θα πρέπει να δούμε τι είναι τελικά αυτά τα ε, διαβατήρια. Ελέγχουν κάθε, κάθε άλλο, όντως οι αρχές. Πρέπει να επανέλθετε και να το ξαναδείτε νομίζω, γιατί η κυρία Πόλσον ε, σωστά μίλησε και μπορώ και να σας στείλω κάποιες ερωτήσεις γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα. Όλοι ξέρουμε ε, ότι ένα από τα προβλήματα είναι το μάκρο της τροφικής αλυσίδας. Και θα πρέπει να πω, Επίτροπε, ότι ο κίνδυνος εδώ είναι ότι ήμασταν εξαιρετικά άνετοι σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Πιστεύετε πως η ΕΦΣΑ αρκεί και τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη όπου οι επιχειρήσεις τους ή μάλλον οι δικοί τους έλεγχοι φαίνονται να είναι τελικά ανεπαρκείς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχήν, η νομοθεσία του χώρα προέλευση δεν προέκυψε έτσι. Προέκυψε εδώ και καιρό. Το νοπό κρέα θα επισημαίνεται από του χρόνου, αλλά η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ήταν αντίθετοι μαζί μου και ε, ακόμα και αν το Κοινοβούλιο συμβουλή, συμφώνησε πως ε, το κρέας μέσα στα μεταποιημένα προϊόντα, τρόφιμα μάλλον, θα πρέπει να σημειώνεται, να σηματοδοτείται. Ε, πρόκειται για μια λυσίδα παροχής που είναι εξαιρετικά περίπλοκη και οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί γιατί θα πρέπει να αναφέρουν τη χώρα προέλευσης. Ε, επειδή πρέπει να το αναφέρουν θα είναι πιο προσεκτικοί, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η εμπιστοσύνη έχει πέσει, οι πωλήσει έχουν μειωθεί για τα έτοιμα γεύματα και είναι το θέμα οικονομικό. Ορισμένοι κατασκευαστές όντως μιλάνε και αναφέρουν την χώρα προέλευσης για το κρέας στα προϊόντα τους και το κάνουν εδώ και πολύ καιρό και γιατί να μην το κάνουν όλοι. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να στηρίξουμε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ ο Ζιλ Πανιό. Μάλιστα Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, είναι απίστευτο η κατάσταση. Με το πρωί έχω μια παράξενη εντύπωση ότι στην ουσία έχετε ε, ε, παραδοθεί κύριε Πίτροπε. Ωστόσο έχουμε να κάνουμε με το πιο μεγάλο σκάνδαλο, τροφικό σκάνδαλο του 20ου αιώνα. Και όταν βλέπουμε τα άλογα, βλέπουμε ότι ταυτόχρονα πρόκειται για το πιο σοβαρό υγειονομικό σκάνδαλο που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Όλοι ξέρουμε ότι τα ζώα και οι αγελάδες ε, είναι φουσκωμένες με αντιβιωτικά και υπάρχουν διάφορα καταστροφικά κοκτέιλ τα οποία πίνουν ε, ή ε, τα ζώα. Ε, μάλιστα σε πρόσφατη έρευνα μιλήσαν για τον συνδυασμό ενός κοκτέιλ που παίρνουν ε, οι αγελάδες που πρόκειται για μικητοκτόνα φάρμακα και τα οποία όταν περάσουν στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο Αλτσχάιμερ. Δεν είναι αστεία αυτά κύριε Επίτροπε. Κάντε κάτι λοιπόν, μιλήστε για τις πολιτικές των κρατών μελών. Θα πρέπει να γίνει μια σπουδαία και ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την καταπολέμηση των ε, διατροφικών σκανδάλων. Ο Σοφοκλής Σοφοκλέους. Τρεις σύντομες διαπιστώσεις τηλεγραφικά. Πρώτον, ορθά αντέδρασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι καταναλωτές και βεβαίως εσείς κύριε Επίτροπε, καθώς και τα κράτη σε αυτό το σκάνδαλο. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια των μέτρων και αποτελεσματικών μέτρων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού. Και η τρίτη Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει καλή νομοθεσία. Η δική μου εκτίμηση, θέση και ερώτηση είναι ότι αυτό που έχετε πει περί αναλογικότητα των ποινών, είμαι από αυτού που πιστεύουν και νομικά ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρότερη εφαρμογή τη νομοθεσίας. Δηλαδή, να το πω απλά και ομά σε αυτό το σκάνδαλο. Καταστολή. Να φοβάται ο πολίτη να φοβάται εκείνο ο οποίο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων μα να προβεί σε τέτοιε ενέργειε και βεβαίω ταυτόχρονα και παράλληλα τα κράτη να λογοδοτούν ενώπιον τη δικαιοσύνη. Σκέφτεστε να προχωρήσετε άμεσα προ αυτή την κατεύθυνση και αν ναι, πώ, πότε και με ποιον τρόπο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επισημάνω και εγώ ότι το πρόβλημα δεν... Μας είπε ότι το πρόβλημα δεν αφήνεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά στην ελληπή άσκηση των ελέγχων από τα κράτη-μέλη. Τι σκοπεύει όμως να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ δεν πιστεύω ότι με την νέα νομοθεσία ή με την ενίσχυση της νομοθεσίας θα αλλάξει η στάση των κρατών μελών ή θα πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι, γιατί αυτό που συνέβη ήδη είναι παράνομο ένα μικρό βήμα μπορούμε να κάνουμε και μία χειρονομία προς τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτό θα είναι παράλληλα με, τους, με το σύστημα ελέγχου να έχουμε και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και για τις απάτες στην επιστηστική αλυσίδα. Η τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική κυρία Γκροστέτ. Η επιχείρηση Φεντής μέσω δοκιμών DNA ε, ανακάλυψε το πρόβλημα. Δεν ε, βρέθηκε το πρόβλημα από τυχαίους ειδικματοληπτικούς ελέγχους των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εξακολουθεί να είναι κλειστή στον χρυσελεφάντινο πύργο της και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ε, των καταναλωτών που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Λένε λοιπόν οι Γερμανοί, θα, εμείς θα καταναλώνουμε μόνο γερμανικά προϊόντα, οι Γάλλοι θα λένε το ίδιο, οπότε πού πάει η εσωτερική αγορά. Είναι σοβαρότατη αυτή η κατάσταση της απόλυσης εμπιστοσύνης και πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλα προβλήματα. Όταν γνωρίζουμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει άδεια για τα ε, ζωάλευρα, για τις χθιοκαλλιέργειες και θα χρησιμοποιηθούν και για, για τους χείρους και τα πουλερικά, τότε είναι που θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότατη κρίση εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων καταναλωτών. Παρόλο που ε, εμεί συμφωνούσαμε τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αντοχή στα αντιβιωτικά, η ελλειπή έλεγχη, η μη συμμόρφωση με τι διατάξει, όλα αυτά συνηγορούν υπέρ τη διαπίστωση ότι έχουμε σοβαρότητα τη παραβιάση εσωτερική αγορά. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε. Έλεγχη, η χνηλασιμότητα, αλλά και η ετικετοθεσία και το περιθώριο που έχει το Κοινοβούλιο, η οικονομική κρίση και βεβαίως ε, κρίση των προπολογισμών. Και όλοι χειροκροτάμε όταν λέμε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αλλά οι ελεγκτές δεν είναι μέρος αυτής της γραφειοκρατίας. Οπότε το ερώτημά μου είναι υπάρχει ε, υπάρχουν στοιχεία της Κομισιόν για το εάν ο αριθμός των ελεγκτών στα κράτη-μέλη. Και τι γίνεται με την ε, ίχνηλασιμότητα αν δεν υπάρχουν ε, επαρκείς ελεγκτές. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε νομίζω αρκετό χρόνο για να απαντήσει ο κύριος Επίτροπος. Πάμε. Ναι, για την τελευταία σας ερώτηση παρά τις δημοσιονομικές περικοπές τις οποίες όλοι περνάμε και η Επιτροπή δεν έχουμε μειώσει τον αριθμό των επιθεωρήσεων των ελέγχων στα κρατή-μέλη. Αυτό συνεχίζεται λοιπόν και θα συνεχιστεί. Αλλά εδώ μπορώ να δεσμευτώ ότι δεν σκοπεύουμε να μειώσουμε τον αριθμό των ελέγχων που γίνονται και αυτό και γιατί βασικά στόχο έχουν ε, τα θέματα ασφάλειας τροφίμων. Θα πρέπει να σας πω ότι με, ε, με ξέπληξε κάπως το σχόλιο του κυρίου Παλμιώζ ότι πρόκειται για, νομικό, για υγειονομικό ζήτημα και άρα και για θέμα ασφάλεια. Αν ήταν θέμα ασφάλεια, όπω είχε γίνει και στο παρελθόν, θα είχαμε προβήσει άμεση δράση Ξέρουμε ότι όταν υπάρχει θέμα ασφάλεια των τροφίμων, ο οικονομικό αντίκτυπο είναι ακόμα χειρότερο. Όταν υπήρχε το θέμα των τρελών αγελάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1% του ΑΕΠ της χώρας ε, ήταν η οικονομική ζημιά. Η Ιαπωνία ε, ήρε μετά από 13 χρόνια την απαγόρευση για το ευρωπαϊκό Κρέα και οι ΙΠΑ ακόμα έχουν την απαγόρευση. 13 χρόνια μετά από το τέλος της ε, ε, Ρώσιας των τρελών αγελάδων. Αφού μου λέτε ότι είμαι άνετος και αυθάριστος, ε, θα σας πρέπει να σας πω ότι δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα και ότι δεν πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει όλα να το τοποθετήσουμε σωστή τους προοπτική. Στους 6.600 τόνους αλόγου αποσύρθηκε, είναι υπερβολικό και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Αλλά είναι ασήμαντο κομμάτι παρόλα αυτά του συνόλου των ε, προϊόντων κρέατος ε, που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην δημιουργούμε λοιπόν και ας μην ε, καλλιεργούμε τον πανικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκομίσουμε διδάγματα, ότι δεν πρέπει να λάβουμε καινούργια μέτρα, ότι θα πρέπει να περάσει, λες και δεν έγινε τίποτα. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αντιθέτως είπα ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε και ανέφερα κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει η Κομισιόν. Επίσης είμαι αντίθετος ε, με την κατηγορία αυτή φυσικά ο θέλει μπορεί να το επαναλάβει ε, αλλά αντι, ε, είμαι αντίθετος με την κατηγορία ότι εμείς δεν αναλάβαμε την ευθύνη μας και τη μοιραστήκαμε θα, θα, το, θα μπορούσατε να το πείτε αν δεν είχαμε κάνει τίποτα αλλά μου είπαν μάλιστα ότι ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση. 8 Φεβρουαρίου η κοινοποίηση, 13 Φεβρουαρίου επίγουσε ε, συνάντηση για τα κράτη που επηρεάζονται, έπειτα πλήρη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, υιοθέτηση ενός ε, σχεδίου παρακολούθησης με κόστος 1 εκατομμύρια ευρώ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια περίοδο ενός μήνα. Εγώ είχα προτείνει τρει μήνες, αλλά τα κρατημέλη προτίμησαν ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης ε, σε άλλους δύο μήνες. Οπότε πάλι θα συγχρηματοδοτήσουμε στο 50% και οι έλεγχοι θα γίνονταν όχι επειδή υπάρχει κρίση ασφάλεια σε τρόφιμα, αλλά για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι πρόκειται για θέμα ασφάλεια. Είναι άδικο λοιπόν να λέτε στην Επιτροπή ότι παρακολουθεί και συγχρηματοδοτεί ελέγχου και θεωρήσει ενώ ταυτόχρονα λέει πως μέχρι τώρα δεν είναι θέμα ασφάλειας. Για, γιατί φυσικά η Κομισιόν θέλει να αποκλείσει τελείω τη δυνατότητα, την πιθανότητα να είναι θέμα ασφάλειας. Γιατί και τα δυο είναι σοβαρά, αλλά το θέμα της κρίσης ασφάλειας τροφίμων, αν αναπτυχθεί, θα ήταν πολύ πιο σοβαρό από ότι ένα θέμα λάθους και ψευδούς ε, επισήμανσης. Οπότε παρακαλώ να με κατανοήσετε, γιατί είμαι αντίθετο σε τέτοιου είδου επικριτικέ που δεν έγιναν εδώ αλλά σε άλλες ότι γιατί κάνετε έλεγχο εφόσον ε, λέτε πως δεν είναι θέμα ασφάλειας των τροφίμων για τις ε, ποινές και τις κυρώσεις. Συμφωνώ με τα όσα είπατε ε, κύριε Ευρωβουλευτές για να φροντίσουμε δηλαδή ότι το, η ποινή να αντιστοιχεί στο έγκλημα και φυσικά θα κάνω την απαραίτητη παραβι... Ε, διαβίβαση προτάσεων στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που μετά θα πρέπει να το εγκρίνουν. Κατά τη γνώμη μου η καλύτερη άποψη θα ήταν να υποχρεώσουμε τα διάφορα νομικά συστήματα των κρατών μελών να ανακτήσουν την ποινή από τα κέρδη τα οποία ε, ήταν αποτέλεσμα της, του, του εγκλήματος. Γιατί αν συνδέσουμε την ε, κύρωση με τα οικονομικά κέρδη που προέκυψαν από την ε, ψευδή επισήμαση, θα έχουμε με μεγαλύτερη αποτροπή από ό,τι τώρα. Σέβομαι βέβαια την αρχή της επικουρικότητας. Μέχρι στιγμής είναι, αποτελεί σημαντικό πυλώνα ε, της ε, Ευρώπης, αλλά όταν ε, αντιμετωπίζουμε κρίσεις, η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει πως αν το κέντρο μπορεί να παρέμβει ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια του τροφίμου, θα πρέπει να παρέμβει. Εάν όχι, θα πρέπει να ασκήσει τις εξουσίες της να επιχρεώσει τα κρατημέλη να προβούν σε ελέγχους μετά από μια κρίση, πέρα από τους τυχαίους ελέγχους που ορίζονται ε, δια νόμου. Και αυτό και προτείνουμε. Όχι, δεν ζούμε λοιπόν σε ε, γυάλινο πύργο παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται, βοηθάμε τα κρατημέλη να βοηθηθούν για την επιβολή της ε, νομοθεσίας αυτής και όσον αφορά τις περαιτέρω εξελίξεις στην νομοθεσία περί σήμανσης, επαναλαμβάνω πως έχω ανοιχτό μυαλό, από όσο γνωρίζω, η Κομισιόν δεν ήταν ε, κατά της αναφοράς της χώρας προέλευσης, τα κρατη ήταν κατά. Ε, ε, και τώρα δεν είμαι κατά. Θα πρέπει να περιμένω το, την εκτίμηση αντικτύπου για να επεκτείνουμε την νομοθεσία περί σήμανσης ώστε να αναφέρεται και η χώρα προέλευσης ακόμα και αν Ορισμένοι λένε ότι αυτό θα αυξήσει το διοικητικό φόρτο των μικρομεσαίων, αλλά πρέπει να κάνουν ότι είναι προς το κοινό συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών και έπειτα. Εάν καταλήξουμε πως αυτό δεν επηρεάζει την ιστορική αγορά, δεν αυξάνει περιβολικά το κόστος και δεν δημιουργεί τεράστιο διοικητικό φόρτο, θα πω, όπως και η κυρία Βίλνοτ, γιατί όχι. Δεν το αποκλείω λοιπόν, απλώ υπογραμμίζω τις δυσκολίες που έχουν ούτως ή άλλως προταθεί και από τα ίδια τα κρατημέλη και από τους ευρωβουλευτές και από τη βιομηχανία και από όλους. Και θέλω να καταστήσω σαφές πως έχουμε διαφορετικές απόψεις για το θέμα, αλλά η Κομισιόν θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο. Και φυσικά θα αποκομίσουμε διδάγματα από αυτήν την υπόθεση τότε θα ζούσαμε σε γυάλινο πύργο αν δεν θέλαμε να αποκομίσουμε τα διδάγματα. Αλλά παρακαλώ τοποθετήστε αυτό το περιστατικό στην σωστέ του διαστάσεις. Παναλαμβάνω ότι είναι σοβαρή παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν πρέπει να... Ε, ε, ότι, ότι να έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποτύχει, ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις τη νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ. Ξέρουμε πως πρέπει να φύγετε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή για τη μία μισή αυτή ώρα. Νομίζω ξεκαθάρισε πως ε, πρέπει να ξανασυζητήσουμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Και ίσως και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα για κάποιες νομοθετικές διαδικασίες να ξανασκεφτούμε τη θέση μας. Και να προσπαθήσουμε να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού μέσω της λογικής διαμόρφωσης ε, του συστήματος της συχνηλασιμότητας και Μπορώ να σας πω πως ε, ε, θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε συναντήσεις με τους ψηφοφόρους μας για να δείτε πραγματικά το τι άποψη έχει ο κόσμος για την ευρωπαϊκή πολιτική τροφίμων είναι συγκλονιστικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που ήρθατε εδώ πέρα και απαντήσατε στις ε, ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ. Ε, λύεται η